Επίτροπε, αρχίζει η συνεδρίαση. Καλή σας μέρα. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Μακάρθη με θέμα εφαρμογή στα κράτη-μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια. Θα ξεκινήσουμε την συζήτηση με την εισηγήτρια. Κυρία Μακάρθη, θα πάρετε το λόγο για τέσσερα λεπτά σας παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κυρία Συγγήτρια. Ε, Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι έχω έξι λεπτά, αλλά θα τα καταφέρω στα τέσσερα λεπτά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και το προσωπικό της Επιτροπής που με βοήθησαν την κατάρτιση της προτάσεως ε, ψηφίσματος για τη διαμεσολάβηση, ε, διότι πρόκειται για μια αναμόρφωση των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών και της νομοθεσίας. Και στην αρχή δεν υπήρχε μια συζήτηση συζήτηση για μια ευρωπαϊκή οδηγία αλλά χρειαζόμαστε στην Ευρώπη ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές για την διαμεσολάβηση και υπάρχουν οικογενειακές διαμάχες σχετικά με την κυδαιμονία, με ε, τα προβλήματα κατοικίας ε, και διάφορα άλλα και η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι δαπανηρή και πολλοί ε, λέγουν ότι ποτέ. Πο, και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω για να μπορέσουν τώρα να έχουν καλύτερη διαδικασία διαμεσολάβησης, να υπάρχει ένα κώδικας συμπεριφοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι βασικό διότι η διαμεσολάβηση έχει αποδείξει ότι υπάρχει ένα 60% ποσοστό επιτυχία στα δικαστήρια, 80% στις διαμεσολαβήσεις αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό ποσοστό των διαδίκων καταλήγουν σε αυτή τη λύση διότι η διαδικασία ε, των δικαστηρίων είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν επιπλέον ε, δικαστικά έξοδα. Ε, αν ήταν το κόστος μίας δίκης για 200.000 ευρώ μακρύ θα ήταν πολύ συντομότερο σε περίπτωση μεσολάβησης και γι' αυτό έχουμε δει ότι οι διαμεσολαβείς στο Ηνωμένο Βασίλειο μπόρεσαν να επιληθούν εντός μίας εβδομάδας μειώνοντας και το κόστος και έτσι επιτρέπουν στους, επιτρέπουν στους διαδίκους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να λύσουν καλύτερα τα προβλήματά τους και ιδίω όταν πρόκειται για τα παιδιά για να μπορέσουν να, καταλάξουν, να καταλήξουν και αυτό είναι σημαντικό και για τις πιέσεις που εξασκούνται μέσα στην οικογένεια για να Φερθώ σε μια άλλη περίπτωση ε, σε μια περίπτωση 10 εκατομμυρίων λιρών με τέσσερις διαδίκους σε τέσσερις διαφορετικές χώρες λύθηκε δια της ε, διαμεσολάβησης σε μια μέρα ε, αφού είχαν ήδη εξοδευτεί 5 εκατομμύρια λίρες για την προετοιμασία που θα χρειαζόταν επιπλέον μια μακριά δικαστική διαδικασία. Προτρέπω λοιπόν εις το να δοθεί αυτή η εναλλακτική λύση επίλυση των νομικών διαφορών και δεδομένων των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να μας στηρίξουν στις περιπτώσεις αυτές διότι υπάρχουν πολλές στην Ισπανία, στην Κύπρο και όπου η διαμεσολάβηση θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιτυχή έκβαση και καταλήγοντας ε, θεωρώ ότι ε, την ε, εποχή που καταρτίστηκε αυτή η διαδικασία μόνο 17 κράτη είχαν κυρώσει την οδηγία του 2008 και συγχαίρω την κυρία Ρέντινγκ που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία παραβιάσεως και ελπίζω ότι θα μπορέσει να υπάρχει μια λογικού κόστους επιτυχής διαδικασία. Αντιπρόεδρος, κυρία Ρέντινγκ. Έχετε το λόγο, Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια, διότι παρουσίασε μια πολύ πλήρη έκθεση για κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι μια θαυμάσια αναλλακτική λύση αντί για ε, δικαστικές διαδικασίες. Όντως η δικαιοσύνη αποτελεί ακρογωνία πλήθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη διαμεσολάβηση όμως έχουμε μια πολύ σημαντική αναλλακτική λύση αντί να πηγαίνουμε στα δικαστήρια όταν έχουμε διασυνοριακές ε, δικαστικές ε, διαδικασίες ή διαφορές. Όπως πολύ σωστά λέει και η συγγήτρια, εξοικονομούμε χρήματα, χρόνο και η διάδικοι ε, ξεπερνάνε τις διαδικασίες πολύ πιο απλά, χωρίς να περνάνε από τραυματικές δικαστικές εμπειρίες. Χρειάζεται βέβαια πολιτική αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο έχει εφαρμοστεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης στις διάφορες χώρες μέχρι τώρα. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι στόχος μας πρέπει να είναι μια ε, αυστηρή εφαρμογή των ε, διατάξεων έτσι όπως προβλέπονται. Μέσα από την έκθεση αυτή πιστεύω ότι περισσότερες χώρες μέλη ακόμα θα επιλέξουν αυτήν την λύση της διαμεσολάβησης γιατί η συγκήτρια έχει δίκιο δεν ισχύει σε όλες τις χώρες μέλη. Δεν υπάρχουν μέτρα δηλαδή που έχουν ήδη προβλεφθεί σε όλες τις χώρες για την οσομάτωση της οδηγίας στην ε, εθνική νομοθεσία. Σε νέες χώρες για παράδειγμα δεν έχει γίνει αυτό καθόλου και πρέπει ακόμα να τεθεί σε εφαρμογή εκεί η οδηγία. Γι' αυτό ακριβώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον Ιούλιο που μας πέρασε διαδικασίες επί παραβάση ε, εναντίον ορισμένων χωρών, των εννέα αυτών χωρών που δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία και έχουν δύο μήνες στη διάθεσή τους για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Θα παρακολουθήσουμε τι θα γίνει με τις εννέα αυτές περιπτώσεις και θα παρακολουθήσουμε επίσης για να δούμε με ποιο τρόπο οι άλλες χώρες μέλη έχουν ήδη εφαρμόσει τις διατάξεις. Θα δούμε κατά πόσο συνάδουν πλήρως με το κείμενο της Επιτροπής και το 2012 σκοπεύω να παρουσιάσω μια ανακοίνωση για τον τρόπο με τον οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία αυτή. Θα επικεντρώνομαι κυρίως τα αποτελέσματα της εφαρμογής της οδηγίας για το κατά πόσο δηλαδή όντως χρησιμοποιείται η διαμεσολάβηση πολύ περισσότερο. Γιατί συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι δεν αρκεί να έχουμε το κείμενο, πρέπει ο κόσμος να το ξέρει ότι υπάρχει η εναλλακτική αυτή λύση και να τη χρησιμοποιεί. Θέλω να προσθέσω επίσης ότι στην οδηγία ε, αυτή ε, η οδηγία αυτή μάλλον δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν ε, στις χώρες τους ε, ανεξαρτήτως από αν πρόκειται για διασυνοριακές διαφορές ή όχι, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την οδηγία, πρέπει να μπορούν και για εσωτερικές ε, διαφορές εφόσον υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την εισηγήτρια και όλους τους ευρωβουλευτές που συνεργάστηκαν. Η πρόταση που έχουμε μπροστά μας βοηθάει πολύ προκειμένου να προωθηθεί η διαμεσολάβηση, να γίνει περισσότερο δημοφιλής και να αντικαταστήσει συχνά δικαστικές διαδικασίες. Τώρα το λόγο θα πάρουν ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Για την ε, κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ο κύριο Ρανχέλ, για δύο λεπτά, παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα βεβαίως να συγχαρώ την κυρία εισηγήτρια γιατί είναι μια πολύ χρήσιμη έκθεση, η οποία θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε πρόοδο στο θέμα αυτό. Έχουμε μια επισκόπηση στην έκθεση της κατάστασης στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας 2008 κάθετος 52 για τη διαμεσολάβηση, σε θέματα εμπορικού δικαίου αλλά και αστικού. Η διαμεσολάβηση είναι μια εξοδικαστική λύση των διενέξεων. Έτσι αποσυμφορούνται τα δικαστήρια. Εξορθολογίζεται το δικαστικό σύστημα εν γέννη. Είναι ένα εργαλείο το οποίο δίνει στους δύο διαδίκους να επιτύχουν μια φιλική λύση, ένα φιλικό διακανονισμό του θέματος ε, με πιο γρήγορους ρυθμούς. Είναι μια λύση λιγότερο δαπανηρή από τη δικαστική διένεξη. Θα πρέπει κανείς να πει ότι έχει μεγάλη σημασία το άρθρο 1 της οδηγίας, να δίδονται κίνητρα δηλαδή στην προσφυγή σε αυτό το μέσο επίλυσης των συγκρούσεων και των διανέξεων. Πρέπει να προωθούνται τα μέσα εξοδικαστικής επίλυσης διενέξεων και θα πρέπει ε, ε, με αυτά να διευκολύνονται ώστε να υπάρχει και καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την πραγματική δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας και δικαιοσύνης. Με τη σημερινή κρίση είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη, αλλά και οι εκπρόσωποι της δικαιοσύνης ε, να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν καλύτερα για τα θέματα αυτά. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, Επίτροπο προσωπικά να ε, προωθήσει μια νομοθετική πρόταση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Γκέριγκερ, για δύο λεπτά επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο την ε, ε, οδηγία και αυτό το υπενθυμίζουμε διότι η εφαρμογή ε, της διαμεσολάβησης δεν είναι ενιαία παντού παρόλο που το Μάιο έληξε η προθεσμία εφαρμογής και ε, μια εναλλακτική ε, λύση για την επίλυση διαφορών μεταξύ των πολιτών μας είναι ε, λογική και μικρού κόστους και βλέπουμε ότι ο χρόνος ο οποίος που καταναλύσκεται για τις ε, ε, για τις ε, διαμεσολαβήσεις είναι από 30 έως 400 ημέρες ενώ είναι πολύ μακρύτερη για τα δικαστήρια. Στην Πολωνία έχει εφαρμοστεί η διαδικασία αυτή και έχουμε ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις αλλά τα στοιχεία της Πολωνίας αποδεικνύουν ότι υπάρχει μόνο ένα μικρό ποσοστό που χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις αυτές ε, για διαμεσολαβήσεις και μόνο 30% των ε, περιπτώσεων επιλύονται δια της ε, διαμεσολαβήσεως ετησίως και πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει στην αρχή του χρόνου δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και γι' αυτό δεν τη χρησιμοποιούν. Πρέπει λοιπόν να προωθηθεί η προβολή αυτής της λύσεως η οποία μειώνει το κόστος, ε, αλαφρώνει το φόρτο εργασίας των δικαστηρίων και επιλύει τα προβλήματα των πολιτών. Γι' αυτό και συγχαίρω την συγγήτρια. Τώρα ε, για την ομάδα των φιλελευθέρων δημοκρατών η κυρία Γουάλης για δύο λεπτά επίσης. Έχετε το λόγο κύριε Γουάλης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και εσά, κυρία Ρέντινγκ για τα όσα είπατε. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό που βλέπουμε το Κοινοβούλιο να εκπονεί έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή. Ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτό το στάδιο τη ζωή της οδηγίας που βρισκόμαστε, συγχρόνω, δηλαδή με τη στιγμή που θέτε σε ισχύ. Και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μακάρθη για το έργο της. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι έδειξε τον καλύτερο εαυτό του εξετάζοντας και κοιτώντας να δει τι γίνεται στις διάφορες χώρες μέλη και εντοπίζοντας τις αδυναμίες, τις ανάγκες αλλά και τα δυνατά σημεία. Θέλω να σας πω ότι και εγώ ήμουν ένας από αυτούς που ήταν πολύ σκεπτικιστές, όπως είπε και η κυρία Μακάρθη. Όντως, όταν προτάθηκε η οδηγία αυτή, είχα τις αμφιβολίες μου, γιατί στην πράσινη βίβλο λέγαμε ότι δεν θέλαμε νομοθεσία γιατί η ανησυχία μας ήταν ότι αποτελούσε απειλή για τις διαφορές και τους πειραματισμούς που λαμβάνουν χώρα όσον αφορά την διαμεσολάβηση στις διάφορες χώρες μέλη. Όμως τελικά με το εργαστήριο με το οποίο ασχοληθήκαμε και με την έκθεση αυτή βλέπουμε ότι καθ' άλλο παρέτσι τα πράγματα. Γιατί οδηγία έκανε καλή δουλειά. Προσέφερε δηλαδή ένα πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει τους πειραματισμούς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τους επιτρέπει να ανθίσουν σε όλες τις χώρες μέλη. Δεν είναι στενός κορσές, όχι, αντίθετα επιτρέπει αρκετή ελευθερία στις χώρες μέλη. Βέβαια δεν λέω ότι όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί, δεν έχουν εφαρμόσει όλες οι χώρες την οδηγία όπως θα έπρεπε, εξακολουθούν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά το απόρριτο για παράδειγμα της διαδικασίας. Όμως νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η διαμεσολάβηση πια θεωρείται μία μέθοδος η οποία είναι πιο σύγχρονη και η οποία επιτρέπει να εφαρμοστεί δικαιοσύνη στις διασυνοριακές υποθέσεις. Ίσως η διαμεσολάβηση να είναι πιο σύγχρονη σήμερα από ότι την εποχή του Μεσαίωνα που θα θυμόσαστε πως λύνονταν ε, τότε παραδοσιακά οι υποθέσεις. Όντως σήμερα αν συγκρίνουμε τη διαμεσολάβηση με τις ε, κλασικές δικαστικές διαδικασίες αυτές οι δεύτερες θυμίζουν Μεσαίωνα. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό για ολόκληρη την κοινωνία. Ευχαριστώ και πάλι την συγκεντρία Εγώ Άλης, και ερχόμαστε στον κατάλογο των άλλων εγγεγραμμένων ομιλητών. Ε, το λόγο θα πάρει ο κύριος Μπαλντασάρε για δύο λεπτά παρακαλώ. Grazie Presidente, gentile commissaria, colleghi e colleghi. Il successo dell'implementazione della direttiva. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η επιτυχία της ε, εφαρμογή της οδηγίας 52-2008 δείχνει ότι η διαμεσολάβηση είναι μια πολύ καλή εναλλακτική λύση στη δικαστική διένεξη, διότι επιτρέπει μια φιλική διευθέτηση των ε, διαφορών και ε, μειώνει το φόρτο εργασίας των δικαστηρίων. Τα κράτη-μέλη ανέλαβαν πρωτοβουλίες, ορισμένα κράτη-μέλη και επιτρέπουν ε, την προσφυγή σε αυτό το μέσο. Ε, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό. Θα ήθελα όμως ε, να σας εφιστήσω την προσοχή σε ορισμένα ζητήματα. Να ακολουθήσουμε καταρχάς το παράδειγμα των κρατών μελών τα οποία ενθάρρυναν τη χρήση αυτού του εργαλείου για εξοικονόμηση πόρων. Θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες τέτοιου είδους δυνατότητες, δηλαδή να γίνουν εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ώστε να ε, αξιοποιηθούν όλα τα εναλλακτικά μέσα για την διευθέτηση των διενέξεων και μάλιστα από πλευράς των επιχειρήσεων. Βεβαίως ε, θα πρέπει εκπρόσωποι της δικαιοσύνης να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτό το ε, σύστημα, να γνωρίζουν και να έχουν συνείδηση της προστιθέμενης αξίας της διαμεσολάβησης, η οποία δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά. Θα ήθελα κι εγώ να τονίσω ότι η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να συμπληρώνει τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως προς το δίκαιο των συμβάσεων μεταξύ άλλων. Δηλαδή η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής θα λειτουργήσει συμπληρωματικά. Όλα αυτά θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε το φόρτο των δικαστηρίων. Λόγο η κυρία Κόνσο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ασχολείται τόσο πολύ με τις εναλλακτικέ λύσεις ε, επιλύσεως των ε, διαφορών διότι είναι δημοκρατικό χαρακτηριστικό και πρέπει οι διαφορές να μπορούν να επιλύονται σε ένα θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουν να υπάρξουν και δεσμεύσεις οι οποίες θα γίνουν σε σεβαστές ιδίως εάν υπήρχε μία διαφορά μεταξύ διαδίκων και πολλές φορές λέγεται ότι αυτό μπορεί να είναι ε, αποτελεσματικό για την περίπτωση της ε, αναλήψεως της κυδαιμονίας των παιδιών και ε, για οικονομικά θέματα ή για συζητήσεις μεταξύ μειονοτήτων που μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να επιληθούν μέσω της διαμεσολάβησης αλλά ε, οι πολίτες δεν γνωρίζουν αρκετά περί τίνος πρόκειται όταν μιλούμε για διαμεσολάβηση και ελπίζουμε ότι η συζήτηση αυτή θα προβάλλει την ε, διαμεσολάβηση και η οποία θα μπορέσει να εφαρμόζεται περισσότερο διότι είναι βασικό ότι είναι στη διάθεση αυτών οι οποίοι διαφορετικά βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση και δεν είναι σε ε, θέση να μπορέσουν να προσφύγουν στο δικαστήριο. Επίσης ε, και το, ο φόρτος εργασίας των δικαστηρίων, η, ε, η δαπάνη για την δικαστική διαδικασία είναι βασικά επιχειρήματα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών σχετικά με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Χρειάζεται μια πιο ενιαία αντιμετώπιση ε, βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη πιστοποίηση και εκπαίδευση των διαμεσολαβητών. Θα έπρεπε τα κράτη να ε, εφαρμόσουν περισσότερες προσπάθειες ε, κατά τρόπον ώστε να μπορέσει κανείς να επιτύχει. Ευχαριστώ. Η κυρία Τέιν. Η ε, εξασφάλιση της εφαρμογής του δικαίου είναι ένα δικαίωμα σε ένα χρόνο ελευθερίας και δικαίου και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ε, δικαιοσύνη είναι επίσης ένα βασικό επιχείρημα και τώρα ο κάθε δικαστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σε κάθε φάση της διαδικασίας να ζητήσει ε, να να προσφύγουν οι διάδικοι σε διαμεσολάβηση για την επίλυση της διαφοράς τους. Ε, δεν υπάρχει ε, πλέον το ε, εμπόδιο της παραγραφής και με την νέα διατύπωση εξασφαλίζεται η ποιότητα και προσπαθούμε να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία αυτή. Έχουν συμμετέχει συμμετάσχει στην προσπάθεια τα περισσότερα κράτη αλλά είναι βασικό να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία αυτή συμβουλευόμενοι εμπειρογνώμονες. Πάρει για δύο λεπτά κυρία Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την δουλειά της ως ε, διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τελικά για τις ε, διεθνείς υποθέσεις που έχουν να κάνουν με απαγωγές ε, παιδιών. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στο σημείο 14, η οποία αναφέρεται στην διαδικασία διαμεσολάβησης και λέει ότι τα διάφορα μέρη μπορούν περισσότερο να λαμβάνουν έτσι υπόψη τη θέση του άλλου και να λύνουν πιο εύκολα τις διαφορές τους. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στους ε, ανθρώπους που έχουν διαφορές μεταξύ τους να εξακολουθούν να έχουν καλές ε, σχέσεις και μετά την επίλυση της διαφοράς. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό όταν εμπλέκονται παιδιά στη μέση. Έτσι μπορεί να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη. Μια τέτοια πρακτική ελπίζω να μπορέσει να επεκταθεί ακόμα περισσότερο και σε όλες τις υποθέσεις τις οικογενειακές μέσα στην Ευρώπη τα μεικτά ζευγάρια αυξάνονται όλο και περισσότερο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 350.000 διασυνοριακοί γάμοι λαμβάνουν χώρα, 150.000 διαζύγια, 20% ε, τα διαζύγια δηλαδή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά που έχουμε ένα διαζύγιο, τα παιδιά μπαίνουν στη μέση και τα χρησιμοποιούν ε, σαν όμοιρους οι γονείς είναι πολλές φορές ο γονιός ο οποίος ε, δεν έχει την κυδαιμονία του παιδιού που όταν έχει το δικαίωμα να δει το παιδί, το παίρνει και το κρατάει και δεν το επιστρέφει μετά πίσω. Τέτοιες υποθέσεις είναι πολλές στην Ευρώπη και μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να βοηθήσει. Τα παιδιά αυτά πολλές φορές μπόρεσαν ε, μέσω της διαμεσολάβησης να ξαναβρούν και τους δύο γονείς τους, να συνεχίσουν να έχουν επαφές και με τους δύο γονείς. Έτσι αποφεύγουμε τραυματικές εμπειρίες για τα παιδιά και επιτρέπουμε και στους γονείς να αντιμετωπίσουν όλα τα οικογενειακά θέματα χωρίς να χρειάζεται να μπουν σε μια δικαστική διαδικασία η οποία τους κοστίζει πολλά και κρατά και πολύ χρόνο. Βλάσακ, για δύο λεπτά επίσης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είμαι πεπισμένος ότι η διαμεσολάβηση και όλοι οι άλλοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης ε, διενέξεων είναι πράγματα εξαιρετικά χρήσιμα και θα ήθελα να τονίσω τα βασικά πλεονεκτήματα. Επίτευξη φιλικής ε, λύσης, ευάρεστης και στα δύο μέρη, ωστόσο υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα. Πρώτον, δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε τα μέρη να πάνε τη διαδικασία μέχρι τέλους. Μετά από τέσσερα χρόνια επίπονων διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν μια οδηγία για τη φιλική διευθέτηση των ε, συγκρούσεων σε διάφορα θέματα εμπορικού δικαίου και αστικού δικαίου. Κατάφεραν λοιπόν να σπάσουν τα ταμπού. Ωστόσο, δεν ε, υπάρχει πλήρης εναρμόνιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η ρύθμιση ε, της διαμεσολάβησης. Ασκείται πίεση στα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους ε, νομοθετικές ρυθμίσεις να τις αποκτήσουν. Το άρθρο 5 προβλέπει υποχρεωτική διαμεσολάβηση, κάτι το οποίο αποτελεί κατάφεωρη αντίφαση με τη φύση της διαμεσολάβησης αυτής καθεαυτής, που είναι μια εθελούσια διαδικασία. εννέα χώρες και η Τσεχία ε, μεταξύ αυτών δεν έχουν ε, υιοθετήσει όλα τα μέτρα που προβλέπονται ε, στην οδηγία. Γιατί αυτό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να γνωρίζουμε μάλλον όλοι ότι οι διαμεσολαβητές στην Τσεχία δραστηριοποιούνται, είναι επιτιδευματίες, λειτουργούν ως σύμβουλοι ε, στο Τσεχικό Κοινοβούλιο συζητήθηκε το θέμα και δεν εγκρίθηκε η θεσμοθέτηση, νομική θεσμοθέτηση της διαμεσολάβησης. Είμαι κατά της υποχρεωτικής εφαρμογής του μέτρου. Ε, τίθενται και άλλα ζητήματα ως προς την ασφάλεια των διαμεσολαβητών αλλά ε, και την δοκιμασία που θα πρέπει να περάσουν για να αποκτήσουν αυτή την ε, ιδιότητα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να τελειοποιηθεί το σύστημα της διαμεσολάβησης σε θέματα που δεν εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο στην Τσεχία. Μένουν δηλαδή ζητήματα εκκρεμή που πρέπει να λυθούν. Ερωτώ λοιπόν, είναι ανάγκη να ασκείται τέτοια πίεση σε ε, κράτη-μέλη που προσπαθούν ούτως ή άλλως. Είστε ακριβείς, διότι πρέπει να φτάσουμε στις ψηφοφορίες 11.30 σήμερα. Είμαστε στη διαδικασία κάτσου διάει τώρα. Έχουν ζητήσει το λόγο τρεις συνάδελφοι. Σας παρακαλώ από ένα λεπτό ο καθένας. Ο κύριος Γιακολίνο πρώτος. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτά που είπε η κυρία Ρέντιν είναι σίγουρα σωστά ε, και ότι ε, το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινοποίηση με μία διαδικασία επιτρέπει σε μια ενιαία αγορά όπως την ευρωπαϊκή αγορά οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να ισχύσουν ενιαία. Είναι βασικός ο ρόλος της ε, δικαιοσύνη, αλλά πρέπει να δούμε και το κόστος της, ε, της διαμεσολάβησης διότι όταν δεν ε, γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων κόστος. Θα πρέπει να γνωρίζει κανείς το κόστος ποιο θα είναι και ε, να έχουμε ε, μεσολαβητές οι οποίοι είναι σωστά κατηρτισμένοι για να μπορέσουν ε, να αποσυμφορήσουν τα δικαστήρια, ιδίω τα αστικά και είναι ουσιαστικό να χρησιμοποιείται για τους ανήλικες αυτή η μέθοδος η οποία είναι πολύ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η επίλυση διαφορών σε εμπορικές δηλαδή διαφορές ή σε προσωπικές διαφορές που έχει αρχίσει από το 2008 σιγά σιγά αρχίζει να αποφέρει καρπούς μέσω της οδηγίας αυτής. Δεν υπάρχουν ε, δυσκολίες. Εκεί όπου χρησιμοποιείται η διαμεσολάβηση διαπιστώνουμε ότι επιτυχάνεται και ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο ό,τι θέλει. Και έτσι μειώνονται οι υποθέσεις που καταλήγουν στα δικαστήρια. Πρέπει να έχει το ίδιο βάρος μια διαμεσολάβηση όπως και μια δικαστική απόφαση. Η διαμεσολάβηση είναι πιο ελκυστική για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα προχωρήσει καλά και θα επεκταθεί στο μέλλον η διαδικασία αυτή. Επίση, στο μέλλον, πέρα από την πρόθεση τη διαμεσολάβηση, πιστεύω ότι θα έπρεπε να ορίσουμε καλύτερα, να εντοπίσουμε καλύτερα την, τις ανάγκες προετοιμασίας των διαμεσολαβητών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Μπρόνς θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι υπέρ ε, της ε, χρησιμοποίησης της εναλλακτικής μεθόδου και επιπλέον είμαι υπέρ ε, του κινήτρου μειώσεως του κούσους, κόστους και να υπάρξουν κυρώσεις για αυτούς που δεν θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν. Δεν νομίζω όμως ότι είναι σωστή η διαδικασία της καταρτήσεως οδηγίας. Τα κράτη-μέρη πρέπει να είναι υπεύθυνα σε τέτοια νομικά θέματα θέματα. Εγώ προτιμώ τη διατησία όπου υπάρχει απόφαση ενώ η διαμεσολάβηση απλώς διευκολύνει την επίλυση αλλά αν όχι αυξάνει το κόστος. Και τέλος ε, πιστεύω ότι σε θέματα οικογενειακού δικαίου είναι ε, σημαντικό ε, και η διαμεσολόβηση και μία διαπραγμάτευση της επιλύσεως είναι καλύτερη. Θα πάρει η κυρία Ρέντινγκ, εξ όνομα της Επιτροπής. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την τόσο καλή δουλειά που έκανε και για τον επικοδομητικό την επικοδομητική συζήτηση και αντικειμενική συζήτηση που μπορέσαμε να έχουμε εδώ στην Ολομέλεια. Όντω, η διαμεσολάβηση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μια σύγχρονη δικαιοσύνη. Όντω, δεν αποτελεί στενό κορσέ για τα κράτη-μέλη. Αποτελεί ένα ευρύ πλαίσιο μέσα στο οποίο τα κράτη-μέλη μπορούν να αναπτύξουν τα δικά του συστήματα. Είναι όμω πολύ σημαντικό για τις περιπτώσεις τις διασυνοριακές διαφορών που είναι συχνά τόσο περίπλοκες και που προσπαθούμε να λύσουμε με ευρωπαϊκά μέσα. Η διαμεσολάβηση είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό για τα ενδιαφερόμενα μέρη, γιατί είναι μια κατάσταση win-win. Όλοι έχουν να κερδίσουν αντί να καταφεύγουν σε τόσο χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Και επιπλέον, όπως υπόθηκε πολλές φορές ε, εδώ, είναι κάτι πολύ θετικό για τις οικογενειακές υποθέσεις που πάνε στα δικαστήρια. Όντω πρέπει να έχουμε μια εκστρατεία ενημέρωση ε, του κοινού έτσι ώστε οι πολίτε να κατανοήσουν ότι μπορούν να προσφεύγουν στη διαμεσολάβηση και πρέπει και να καταρτήσουμε του διαμεσολαβητέ ώστε να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά του κάθε φορά που αναλαμβάνουν μια διαμεσολάβηση. Με ρωτήσατε και διάφορα πράγματα, κυρία Πρόεδρε, για την ε, εναλλακτική διαμεσολάβηση του NDR. Θέλω εδώ να ενημερώσω το Σώμα ότι το Μάρτιο του 2011 ε, έγινε η διαβούλευση με το κοινό όσον αφορά τις εμπορικές ε, συναλλαγές και οι απαντήσεις που πήραμε δείχνουν ότι στηρίζονται τα προγράμματα αυτά σε περιπτώσεις εμπορικών διαφορών και διαφορών με τους καταναλωτές. Ο Επίτροπος Νταλίος, συνάδελφό μου, μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα ετοιμάσει μια νομοθετική πρόταση για το ADR και μετά στα πλαίσια της ψηφιακής ατζέντα το 2012 θα υπάρξει μια ρύθμιση για online ADR. Εγώ η ίδια ζήτησα από τις υπηρεσίες μου να εξετάσουν το θέμα του ADR ε, στη, για τις περιπτώσεις δηλαδή σχέσεων επιχειρήσεων με επιχειρήσεων και προβλέπεται σχετική νομοθεσία μέσα στο 2012. Και επειδή εκφράσατε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις οικογενειακές υποθέσεις και διαφορές, θέλω να σας πω ότι προκειμένου να δώσουμε συνέχεια στην υπουργική διάσκεψη που έγινε για την οικογενειακή διαμεσολάβηση υπό τη Βελγική Προεδρία το Δεκέμβριο του 2010 και τις συζητήσεις που ακολούθησαν στο Συμβούλιο, ξεκίνησε μια ομάδα εργασίας για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακά ζητήματα. Βλέπετε δηλαδή ότι παίρνουμε τα θέματα αυτά πάρα πολύ σημαντικά και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί πολύ σωστά είπατε, για τα παιδιά η διαμεσολάβηση είναι πάντα μια πολύ καλύτερη λύση από ότι μια δικαστική διαδικασία. Πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Το, η εισηγήτρια θα κλείσει τη συζήτηση. Έχετε δύο λεπτά κυρία Μακάρθη. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Για να απαντήσω στον κύριο Μπρόντς, να πω ότι σαφέστατα δεν έχετε καμία ιδέα πόσες πολλές διασυνεροϊκές διανέξεις ε, ταλανίζουν τους, τα μέλη της περιφέρειάς τους της περιφέρειάς σας. Νομίζω ότι μιλάτε βάσει ιδεολογίας. Οι πολίτες εποφελούνται από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έρθετε σε επαφή με διαμεσολαβητές από το Ηνωμένο Βασίλειο για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι αυτά που κάνουμε εδώ. Θέλω να πω στην κυρία Ρέντιν ότι προσδοκούμε με αγωνία την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ADR. Και θέλω να τονίσω αυτό το οποίο είπε και η κυρία Wallis οφείλουμε να διατηρήσουμε την, ε, τις διαφορές και την ποικιλότητα, αν θέλετε, μεταξύ των διαφορών χωρών μελών, ε, να μιλήσουν τα κράτη-μέλη με τους επαγγελματίες διαμεσολαβητές, με τους ειδικού, με τους αρμόδιους φορείς, γνωρίζουν ποιο είναι το καλύτερο, ώστε ε, να έχουν οι πολίτες μας καλύτερη πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Και η Επίτροπος θα πρέπει να το κάνει αυτό. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι